Λοιπόν και τα δικαιώματα των γυναικών. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην ε, Τουρκία για την επίσημη επίσκεψη. Ε, το Κοινοβούλιο, συναντήθηκα με εκπροσώπους της κοινωνίας ε, των πολιτών, ε, μίλησα με τον ε, Πατριάρχη Βαρθολομέ για την κατάσταση των χριστιανών στην Τουρκία. Θέλουμε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση, ενθαρρύνοντας την τουρκική πλευρά να υιοθετήσει μια θετική προσέγγιση για να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα πρόβλημα εν ώψη και τη ε, επερχόμενη Κυπριακή προεδρία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε θέματα όπως ε, δικαιώματα των μειονοτήτων, δικαιώματα των γυναικών και... Ε, τους ενημέρωσα ότι λίαν Συντόμος ε, θα αρχίσουμε τις εργασίες μας σχετικά με την αντιμετώπιση της ε, κρίσης ε, μετά την ε, έκπτωση του κυρίου Μουμπάρακα στην Αίγυπτο διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση, οι αρχές, ε, τα πολιτικά κόμματα καθώς και η κοινωνία των πολιτών ε, θα πρέπει να συνεργαστούν ε, και να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή του λαού, η λαϊκή εντολή μετά τις εκλογές. Επίσης έχουμε γενικές κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μαρόκο μετά τις μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο θα έχει διευρυμένες εξουσίες, περισσότερες αρμοδιότητες Ε, το ίδιο ισχύει και για την κοινοβουλευτική συνέλευση της ε, Αιγύπτου. Δυστυχώς ε, η αποστολή παρατήρησης των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε αποδεκτή στο Μαρόκο. Λυπούμεθα γι' αυτό. Ε, υπάρχουν διάφορες αιστείες έντασης ε, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, όπως όλοι γνωρίζετε. Ε, δείχνουμε ιδιαίτερη κατανόηση και συμπόνια για τους νότιους γείτονές μας. Θα ήθελα να περάσω τώρα στις επίσημες ανακοινώσεις. Informuję, że zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 i 4 regulaminu Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της του εσωτερικού κανονισμού 3 ε, και 4 του εσωτερικού κανονισμού έχει, έχει ε, επικυρωθεί ότι ε, ζήτησε επικύρωση της θητείας του ο Ευρωβουλευτής Κέντ Γιώχανσον από τις